να σας ζητήσω να συζητήσουμε νωρίτερα τα θέματα της απόψινής βραδιάς στις 8. Ωραία, εγκρίνεται η τροποποίηση. La seduta è sospesa. Αναβάλλεται η σύνοδος μέχρι τις 8. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.